Πρόκειται για προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδιαμετρότητα. Για να ξεκινήσουμε θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Αρένα, συντάκτρια της ερώτησης αυτής. Merci, euh, Monsieur le Président. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία συζήτηση που κάναμε εδώ στην Ολομέλεια για την άδεια μητρότητας ε, έγινε τον Ιούλιο του 2014. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και από τότε δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα θα έλεγε κανείς. Ε, κι όμως έχουν γίνει ορισμένα πράγματα. Ο Φρανς Τιμέρμανς θέλει να ανακαλέσει την οδηγία ε, για την άδεια μητρότητα. Το Συμβούλιο κάνει ότι δεν ακούει και εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο. Πρέπει και εμείς, ε, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα μία ακόμη φορά να καταγγείλω την αδράνεια του Συμβουλίου, όπως επίσης και το προηγούμενο που σημαίνει κάτι τέτοιο. Ε, δύο όργανα συμφωνούν, αλλά το Συμβούλιο ε, δεν τοποθετείται ή μάλλον τοποθετείται πολύ διαφορετικά από τα άλλα δύο όργανα. Είναι κάτι το απαράδεκτο και σε θεσμικό επίπεδο. Δεν σέβεται τα δύο άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης και απαράδεκτο ε, για τα εκατομμύρια μητέρες και παιδιά ε, που δεν ε, μπορούμε να τους εγγυηθούμε κοινωνική δικαιοσύνη δεν ε, σημαίνει ότι αν κανείς ε, πετάξει στα σκουπίδια την ε, οδηγία για την μητρότητα θα πετύχουμε τους στόχους που εξήγηλε ο κύριος Γιούνκερ γιατί ουσιαστικά πολλές γυναίκες είναι σαν να τιμωρούνται επειδή γίνονται μητέρες και τι θα απογίνουμε εάν το να κάνει κανείς ένα παιδί σημαίνει φτώχεια. Το ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο ε, δι, ε, θέλει η Ευρώπη να είναι μια πραγματική ε, Ευρώπη 3α ε, από απόψεις κοινωνικής δικαιοσύνης γιατί το 1992 είναι η πρώτη ημερομηνία για την πρώτη οδεία μητρότητα δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα τώρα βρισκόμαστε στο 2015 λέγαμε σήμερα το πρωί ότι αν πρέπει η Ευρώπη 20 χρόνια για να νομοθετήσει για κάτι δεν θα πάει πουθενά, ειδικότερο όταν πρόκειται για κοινωνική νομοθεσία. Αυτό λοιπόν που λέμε στο Συμβούλιο, αυτό που λέμε στην Επιτροπή, αυτό που λέμε και εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ότι αυτές οι γυναίκες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Πρέπει να μπορούν να συμφιλιώσουν επαγγελματικό και οικογενειακό βίο. Δεν είναι δυνατόν να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ τη μητρότητα και της ε, καριέρα του. Πρέπει να μπορούν ε, να ε, διεκπαιρεώσουν όλους του τους και ω μητέρες και ως επαγγελματίες δεν πρέπει να είναι θύματα ε, του pension pay gap, ε, της διαφοράς και στις αμοιβέ και στην συνταξιοδότηση, γιατί είναι μητέρες, ε, γιατί κινδυνεύουν κάποια μέρα, και αυτό ακούμε σήμερα, κινδυνεύουν να γίνουν μητέρες. Φαντάζεστε στην Ευρώπη είναι δυνατόν να είναι κανείς, να αποτελεί ένα κίνδυνο για να, το να γίνει κανείς μητέρα, ένας κίνδυνος ε, για ε, ε, την κοινωνία. Μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Γι' αυτό ακριβώς που ζητούμε, αυτό ακριβώς που ζητούμε σε αυτό το ψήφισμα είναι όλα αυτά να σταματήσουν να υπάρχουν. Οι γυναίκες αυτές, ε, οι μητέρες ε, όσες βρίσκονται σε άδεια μητρότητας να μπορούν να ε, αμείβονται σωστά για να μην βρίσκονται στη φτώχεια, να μπορούν να αναλάβουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, να μπορούν να διεκπαιρεώσουν το ρόλο τους γυναίκες, μητέρες και εργαζόμενες και να έχουν μια αξιοπρεπή θέση στην κοινωνία μας. Κύριε Επίτροπε, ξέρω ότι σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και ότι ε, συμμετέχετε ενεργά. Σας ζητώ να μην περιμένουμε άλλα 10 χρόνια για να μπορέσουμε να δώσουμε ε, τη δυνατότητα αυτή σε αυτές τις Ευρωπαίες μητέρες. Ε, βασίζομαι και σε εσά και στο Συμβούλιο. Όλη την ώρα το επαναλαμβάνουμε, ε, συνεχώς λέμε στο Συμβούλιο ότι είναι αυτό που ζητούμε. Ας προσπαθήσουμε να συνασπιστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να γίνουν σεβαστές αυτές οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Λουκαντσίτσιλ από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη, κύριε Επιτρόπε. Να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την πρόταση τη Κομισιόν για αναθεώρηση τη οδηγία ε, περί αδεία μητρότητα. Του τελευταίου μήνε η Προεδρία έχει συναντήθει με το εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου σε πολλέ περιστάσει για να συζητήσει το θέμα αυτό. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αποσύρει την πρόταση εάν δεν σημειωθεί εφικτή αυτή η πρόοδος μέχρι το καλοκαίρι στις διαπραγματεύσεις. Θα υπάρξω ειλικρινής μαζί σας. Η πρόταση ως έχει σαφώς δεν την χάνει υποστήριξη το Συμβούλιο. Η θέση του Συμβουλίου δεν αφήνει περιθώριο για περαιτέρω ελιγμούς. Πρέπει να είμαστε επίσης ρεαλιστικοί όσον αφορά το εξή. Η θέση του Κοινοβουλίου και οι προσδοκίες του από το αρχείο αυτό διαφέρουν σημαντικά από τις προσδοκίες ε, του Συμβουλίου. Σεβόμαστε τη θέση αυτή. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση όπως έχει σήμερα δεν θα μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο στο αρχείο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αξιότιμα μέλη, Επιτρέψτε μου να τονίσω ένα πράγμα. Η θέση του Συμβουλίου δεν ήταν ε, κάτι που αποφασίστηκε απλά. Βασίστηκε σε πολύπλοκη σκέψη. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες. Αφιερώθηκε εξαιρετική καλή βούληση από τις προηγούμενες ε, προεδρίες. Η Προεδρία δεν μπορεί να δραμώνει της. Δεσμεύεται από τη Βούληση των Κρατών Μελών ακριβώς όπως και το Κοινοβούλιο δεσμεύεται από τις απόψεις των μελών του. Παρά τις δυσκολίες που χαρακτήρισαν ε, αυτό το αρχείο, αυτό το θέμα, θεωρώ ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο παραμένουν ενωμένα στη δέσμευσή τους προς τις γυναίκες της Ευρώπης και προς τις εργαζόμενες μητέρες ειδικότερα. Το Συμβουλίο επανειλημμένως έχει τονίσει τη σπουδαιότητα που έχει το να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τους άντρες στον αγώνα συμφιλίωσης της ε, ε, επαγγελματική ε, και οικιακής ζωής και οικογενειακής ζωής. Η πρόθεση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας δεν αποτελεί απλά θέμα ισότητας. Είναι και ένα σημαντικός παράγον ο οποίος συμβάλλει στην συνολική οικονομική ανάπτυξη. Με αυτό το γενικότερο στόχο υπόψη, μετά από 7 έτη προσπαθειών, άκαρπων, θα θέλαμε να δούμε μια νέα αρχή, μια νέα φετηρία για αυτό το θέμα. Μια νέα πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει καλύτερη βάση για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο ώστε να συνεργαστούν από κοινού για να βελτιώσουν τις ε, συνθήκες συμφιλίωσης της ε, επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για άνδρες και γυναίκες. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την προστασία των εγγύων και των γαλλουχουσών εργαζομένων. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταφέρει να συμμεριστεί τις απόψεις του Συμβουλίου ε, ότι υπάρχει ανάγκη να υιοθετήσουμε μια πιο ε, διορατική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Υφυπουργέ. Και τώρα η Επίτροπος ε, κυρία Ζουρόβα εξ ονόματος της Επιτροπής. Ε, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την εμπλοκή της και τις προσπάθειες που κατέβαλε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της ε, οδηγίας όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε άδεια μητρότητας. Επίσης και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς της κυρίας Γαρθία Πέρες για να εξευρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Δεσμεύεται στεναρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Αναγνωρίζει την ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να μπορούν να συμφιλιώσουν την εργασιακή τους ζωή και να μπορέσει να συνδυαστεί αυτή με την οικογενειακή τους ζωή. Έχει τονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα ότι είναι πρόθυμη να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου πλάκι μέσα σε διαρκείς προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και η Προεδρία ΕΝΗΝ και οι προηγούμενοι εργάστηκαν στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας λύσης. Χάρη στην κυρία Αρένα υπήρχε η δυνατότητα, υπήρξε η δυνατότητα να ανοιχνευθούν νέες δυνατότητες ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα των άμοιβων, πράγμα το οποίο αποτελούσε θέμα τριβής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκόλυνε άτυπες συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ήταν πάντα υπέρ των συγκεκριμένων συζητήσεων και χειροπιαστών αναλύσεων με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσει να υπάρξει κίνηση προς μια συμφωνία. Και επανέρχεται το θέμα τώρα, η συζήτηση ε, στο Συμβούλιο με βάση τις προτάσεις ε, των εισηγητών για να μπορέσει να αποτροχοπεδηθεί η κατάσταση που αυτή τη στιγμή έχει παγώσει και έτσι να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε την προθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη θέση του και την προθυμία να σημειωθεί πρόοδος. Δυστυχώς, μια ολόκληρη ομάδα κρατών μελών είναι αντίθετη στην προώθηση των διαπραγματεύσεων επ' αυτού του χαρτοφυλακίου. Συμφωνώ πολύ ότι υπάρχει, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα, ωστόσο δεν έχουν πιστεί ότι αυτή η πρόταση η οποία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια δεν θεωρούν ότι θα, επιλύ, δεν θεωρούν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα τα οποία υφίστανται. Υπάρχει παρόλα αυτά μια τάση προς μια νέα εκκίνηση από πλευρά Συμβουλίου. Εξακολουθούμε να είμαστε πρόθυμοι στο να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση με τους συνομοθέτες. Όπως έχουν τώρα όμως τα πράγματα δεν βλέπει κάποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεκκλίνει από τις δικές της θέσεις στο πρόγραμμα εργασίας να αποσυρθεί δηλαδή αυτή η πρόταση και να αντικατασταθεί με μια άλλη αν δεν εξευρεθεί δηλαδή μια συμφωνία μετά από 6 μήνες. Τώρα μια νέα κίνηση από μηδενικού σημείου φαίνεται να είναι η καλύτερη ε, γραμμή πορείας και θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να δει την κατάσταση, να επανεξετάσει την κατάσταση των εργαζομένων γονέων είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε μια νέα πρόταση με ένα νέο ξεκίνημα. Γνωρίζουμε ότι κυρίως οι γυναίκες είναι εκείνες που πλήττονται από αυτό που αποκαλούν οι οικονομολόγοι την ποινή της κυρώσης της μητρότητας. Οι δυνατότητες να συμμετέχουν οι γυναίκες ε, όταν γίνονται μητέρες στην αγορά εργασίας ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Επίσης το θέμα των πληρωμών των αμοιβών και να δούμε και το ποσοστό που παραμένει σε 16% και το, τις διαφορές και τις μισθολογικές και τις συνταξιοδοτικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα δημογραφικής συρρήκνωσης. Υπάρχουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά και δημοσιονομικά προβλήματα τα οποία συνδέονται λόγω αυτής της κατάστασης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει η Ευρώπη να κάνει χρήση όλων όλων των ε, ικανοτήτων και όλου του δυναμικού που υπάρχει. Οι γυναίκες έχουν καλύτερα προσόντα από ό,τι οποτεδήποτε στο παρελθόν. Έχουν δεξιότητες και ικανότητες περισσότερες από τους άντρες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αμελούμε και να αγνοούμε αυτά τα προσόντα των γυναικών. Όταν υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστικότητα παγκόσμια και η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, πρέπει να υπάρξει μια πιο ισοσταθμισμένη κατάσταση ώστε να μπορούν γυναίκες και άντρες να ιδρύουν συνεδρίου τις οικογένειες που επιθυμούν. Πρέπει να υπάρχει επιλογή για τα ζευγάρια. Πρέπει επίσης και οι άντρες να μπορούν να έρθουν στο ύψος των υποχρεώσεών τους. Πολλοί άντρες θα ήθελαν να αναλώνουν να παίρνουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν μια σωστή εξισορρόπηση εργασιακού βίου και ιδιωτικού οικογενειακού βίου. Αυτό θα βοηθήσει και την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και θα προαγάγει την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα. Οι προκλήσεις των εργαζομένων γονέων ξεκινούν με την άφηξη ενός νέου παιδιού, ενός μωρού. Δεν σταματούν όμως εκεί. Πρέπει να υπάρχουν και περιθώρια ελαστικότητας και ευελιξίας. Πρέπει να υπάρχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διασφάλισης ε, των, της φροντίδας των παιδιών, ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα επιλογής ε, που θα έχει νόημα για τους ανθρώπους. Καθώς επίσης και η μέρημνα των ηλικιωμένων και όσων εξαρτώνται από, την, από τις οικογένειες σήμερα. Όλα αυτά να γίνονται όμως με έναν ευφυή τρόπο, με ένα εφάνταστο ευφυή τρόπο ώστε να μην αποτύχουν ή και να μην οδηγήσουν σε προβλήματα. Για αυτούς τους λόγους ε, στοχεύω στο να εξετάσω αυτό το θέμα όπως και με τους συναδέλφους μου Ντομπρόφσκης και την κυρία Τάισεν και να δούμε το πλαίσιο, το ρυθμιστικό που μπορεί να βελτιωθεί, να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η θέση και των γυναικών στις κοινωνίες και στις επιχειρήσεις και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκε του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πάντα σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορεί να προβληματιστεί από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο για όλε τι πτυχέ που πρέπει να καλυφθούν και να ληφθούν υπόψη. Θα γίνει και μια δημόσια διαβούλευση και θα συμβουλευτούμε με του κοινωνικού εταίρου με τι καλύτερε οδού και τρόπου στο πεδίο των κοινωνικών πολιτικών όπω προβλέπει και η συνθήκη θα εξεταστούν σε πλήρη εμβέλεια τα μέτρα που μπορούν να αναλυθούν και τα, οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να είναι οι πιο αποτελεσματικές. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, προσβλέπω στο να ακούσω τις απόψεις σας και βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ζαμπόρσκα Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μιλάμε σήμερα για την οδηγία σε σχέση με την αδιαμητρότητα και όχι μόνο μιλάμε για ένα έγγραφο που αφορά την προστασία της υγείας και τις θέσεις εργασίας ε, για τις ε, ε, εγκυμονούσες τα κράτη πρέπει να προσφέρουν σήμερα 14 εβδομάδες ε, αδιαμητρότητα. δύο εβδομάδες είναι υποχρεωτικές, ωστόσο οι γυναίκες ε, διατηρούν, πρέπει να διατηρούν τη θέση εργασία τους και να διατηρούν και κάποιο βασικό εισόδημα, ίσως όχι ολόκληρο. Αυτό αναφέρεται στην οδηγία του 92 που ισχύει ακόμα σήμερα. Στο μεταξύ η Κομισιόν ε, προετοίμασε μία αναθεώρηση, το Κοινοβούλιο έλαβε θέση, αλλά το Συμβούλιο δεν θέλει να διαπραγματευτεί τη θέση αυτή. Όσον αφορά την οδηγία που αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας για τις γυναίκες, αυτή μεταμορφώθηκε σε ένα μέσο το οποίο αφορά και την ισότητα των φύλων, αλλά μπλοκαρίστηκε στο Συμβούλιο και οι γυναίκες έπεσαν θύματα των πολιτικών φιλοδοξιών. Η παράταση ε, τη ένδυση μητρότητα σε 18, 18 εβδομάδες όπως προβλέπεται διεθνώς θεωρώ ότι αυτέ οι γυναίκε που παραμένουν στο σπίτι πρέπει να λαμβάνουν πλήρες, ε, πλήρω, τον πλήρη μισθό τους. Με απογοητεύει ότι αυτό που ζητείτε και το γεγονό ότι ζητάμε από το Συμβούλιο να ξαναμπεί σε διαπραγματεύσεις ε, επί ενό αντικειμένου που περιλαμβάνει σφάλματα. Μιλάμε για βελτίωση των συνθηκών εργασία για τι έγκυε γυναίκε, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη τη δική του οικογενειακή πολιτική. Ω η ηγέτρια του ΕΛΚ πρέπει να πω ότι αν αυτό το ψήφισμα εγκριθεί ω έχει, οι συνάδελφοί μου θα απέχουν από την ψηφοφορία. Όσκα, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Φρουντζουλίκα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ κύριε Φρουντζουλίκα. Yeah, it's okay.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 Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ήσασταν σκιώδη συζυγήτρια, μήπως ε, νομίζετε ότι είναι επιτέλους η στιγμή για το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις ε, για την οδηγία, για την άδεια μητρότητας με το Κοινοβούλιο και να λάβει την ευθύνη για την άρνηση ε, όλων αυτών των βελτιώσεων για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, των γυναικών που είναι σε άδεια μητρότητας ή ε, που είναι λεχόνες και θυλάζουν. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπατε. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να ξαναμπεί στη διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των ε, εγγύων και των γαλουχουσών και των λεχόνων. Πρέπει λοιπόν να, ε, να σεβαστούμε, να τηρήσουμε την οδηγία αυτή που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Λόπες. Bien, el Consejo... Μάλιστα, το Συμβούλιο είπε ότι θα ομιλήσει ειλικρινά και ευθέως και θα το κάνουμε και εμείς και να δούμε τι συνέβη εδώ. Το Συμβούλιο και η τρέχουσα Προεδρία αποφάσισε από την πρώτη στιγμή να καταποντήσει αυτή την πρόταση, αυτή την οδηγία. Όταν γίνεται λόγος για το Κοινοβούλιο λέγεται από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε ελαστικοί, ευέλικτοι και να διαπραγματεύσουμε. Έχουμε μια παλαιά πρόταση και θέλουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο όμως δεν ανταποκρίθηκε με κανένα τρόπο από και επιπλέον πρόκειται για μια οδηγία, για μια οδηγία ισότητας προφανώς, ισότητας των φύλων και που αφορά μέσα την εργασιακή αγορά και τη δημογραφική μας κατάσταση και τις προκλήσεις μας και θα έπρεπε να αποτελεί τμήμα της ανάκαμψης, της οικονομικής ανάκαμψης. Και το χειρότερο, κάποιοι από το Συμβούλιο δεν με παραξενεύουν καθόλου με τη στάση τους. Οι γυναίκες είναι γνωστό ότι έχουν μικρότερες συντάξεις επειδή εθελοντικά, λέει, δεν εργάζονται για να έχουν παιδιά. Αυτό είπαν και δεν με παραξενεύει καθόλου το ότι έχουν μια τέτοια θέση και τοποθετούνται έτσι ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο για την ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκέρλινγκ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συναδελφοί. Δεν είναι σύμπτωση ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία για τις έγκες εργαζομένους και τις καλοχούσες και τις λεχόνες ε, έχει γίνει γνωστή ως οδηγία για την αδιαμητρότητα. Δεν είναι απλά για γλωσσικούς λόγους. Έχει ε, μεταμορφωθεί ε, λόγω της οδηγίας για την ίση πληρωμή. Τίθε θέμα εδώ επικουρικότητας και έχει έρθει ώρα η Κομισιόν να την αποσύρει. με όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται ανώτητο και αυτή η προφορική ερώτηση τονίζει αυτό το σημείο. Αν το Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει με την αρχική πρόταση όπως ε, γίνεται με τις, ε, ε, σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα είχαν επιτευχθεί όλα αυτά πριν από πέντε χρόνια. Το ότι έχουν πεισμώσει ορισμένα μέλη είναι η αιτία που έχει καθυστερήσει η πρόοδο. Προτείνω λοιπόν η Κομισιόν να αποσύρει αυτή την πρόταση και να πάψει να χάνει χρόνο με αυτό το θέμα. Ε, έχετε μια μπλε κάρτα. Έχετε, κυρία Γκέρλιν, μια μπλε κάρτα από την κυρία Αρένα. Τη δέχεστε? Παρακαλώ. Ήθελα απλά να κάνω μια ερώτηση λέει στην ε, κυρία Γκέρλινγκ. Η άδεια μητρότητα ε, και η σχετική οδηγία υπάρχει από το 1992. Αφορά την προστασία των γυναικών στο χώρο εργασία, Είναι λοιπόν μια οδηγία περί της υγείας ε, γυναικών εγγύων, γαλουχουσών και λεχόνων. Υπάρχει από το 1992 η οδηγία που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια αναθεώρηση της οδηγίας του 92. Όταν εσείς μιλάτε λοιπόν για επικουρικότητα, σε τι αναφέρεστε. Αφού από το 1992 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει τέτοια μέτρα. Ε, well, presumably the... Το ερώτημα αφορά την κατανόησή μου της οδηγίας. Δεν ήταν ουσιαστικά ερώτημα, αλλά να σας πω το εξής. Είναι σαφέστατο ότι η πρόταση αναδιατύπωσης ε, έχει προσκρούει στην ε, επικουρικότητα και ε, επιθυμεί να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που είναι ε, λογικό να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη της ομάδας μας, η άδεια μητρότητας είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να προωθούνται τα δικαιώματα των γυναικών. Το θέμα είναι ε, όλες αυτές, ε, οι, όλα, όλα αυτά τα ζητήματα που τίθενται χωρίς καμία απολύτως ευελιξία, αν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν έξι. Η κυρία Μπεθέρα Μπαστερετσέα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε Γιώροβα, κυρία Κανίνα θυμόσαστε τι συνέβαινε το 1992. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, διότι την επόμενη χρονιά γεννήθηκε ο γιος μου και μου άλλαξε η ζωή και το θυμάμαι πολύ καλά. Όλη η κοινωνία άλλαξε, οι γυναίκες, η οικονομική κατάσταση, η Ευρώπη των 28 δεν μπορεί να έχει μια οδηγία της Ευρώπης των 12 κρατών μελών. Είναι ευθύνη μας και πρέπει να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας και να δώσουμε κάτι το οποίο θα δίνει λύσεις στις ανάγκες τους εκείνο το οποίο του ανησυχεί. Άλλε χώρε γύρω μα έχουν αντιδράσει και έχουν υιοθετήσει ρυθμίσει που βελτιώνουν τα συστήματα, δίνουν μεγαλύτερα δικαιώματα, μεγαλύτερη προστασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σε θέση εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια να εγκρίνει μια πρόταση για αυτή την γονεϊκή άδεια που ήταν πιο φιλόδοξη από εκείνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έγινε με το Συμβούλιο. Σε αυτά τα πέντε χρόνια ούτε μια λέξη, απόλυτη σιωπή, ούτε μια πρόταση δεν τοποθετήθηκε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο θέμα. Μία τροχοπέδηση απόλυτη και συστηματική. Παραβιάζεται η αρχή της συναπόφασης των συνθήκων. Και εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού και σε σχέση με το Συμβούλιο ζητούμε ευθύνη, υπευθυνότητα, διοργανική και διαθεσμική υπευθυνότητα και πνεύμα υπέρ της Ευρώπης και ζητούμε να γίνει κάτι παραπάνω από ένα παθητικό ρόλο. Δεν μπορεί να απορριφθεί αυθαίρετα μια πρόταση που είναι αναγκαία. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα αναγκαία κριτήρια. Εγώ πιστεύω ότι ομιλώ εξ ονόματος των συναδέλφων όταν σας λέω όταν σας λέω ότι είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε <clears throat> και αν υπάρξει νέα εκκίνηση όπως λέει η κυρία Ζούροβας πείτε μας πότε να γίνει αυτό ανταποκρινόμενοι σε σχέση με την εντολή που έχουμε από τους ε, πολίτες μας, ε, μεταφέροντας τις προτάσεις ε, και τις ανησυχίες τους. Ευχαριστώ. Για την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς, το λόγο έχει η κυρία Ζούμπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα από αυτά τα θέματα που ιδιαίτερα καταδεικνύει την φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφάσεις για μισθολογικές περικοπές. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει συμφωνία επ' αυτού οι χώρες που είναι όμοιροι των τραπεζών, των επιχειρήσεων και πάλι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, σε σχέση με τα πλοία για την Λιβύη και η αντιμετώπιση τους συμφωνούν. Τώρα, για τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών και ε, ένα ελάχιστο διάστημα πληρωμένων ε, ε, διακοπών για τις γυναίκες μητέρες περιμένουμε, περιμένουμε και δεν υπάρχει συμφωνία ενώ θα έπρεπε να υπάρχει οπωσδήποτε να ευδοκιμήσει και όπως είπε η Επίτροπος επιθυμούσε να υπάρξει λύση όμως είναι πολιτική βούληση και λύση και δεν είναι διοικητικό το θέμα και πρέπει να υπάρξει υποστήριξη και όταν λέει η κυρία Επίτροπος ότι είναι, υπάρχει η προθυμία για μια νέα κίνηση. Τι σημαίνει αυτή η νέα κίνηση το νέο ξεκίνημα. Σε σχέση με την πρόταση που είχε ε, ζητηθεί από το Συμβούλιο, νέα κίνηση τι σημαίνει. Μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ε, γυναικών. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι οπισθοδρόμηση σε σχέση με την θέση που είχε υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά τα άλλα <clears throat> που λένε ότι είναι ακριβώς ε, δημοκρατικό ζήτημα. Δεν είναι όμως θέμα δημοκρατικότητας εδώ. Διότι όταν βλέπουμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα δικαιώματα, δεν είμαστε εμεί που κρίνουμε γι' αυτό και θέλουν οι εργαζόμενε να έχουν ε, το πλαίσιο που να διασφαλίζει τα δικαιώματά του και όχι να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και να ε, μην λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματά του. ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Φάνα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Για τους πρασίνους θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία από πλευρά Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αδιανόητη η προαναγγελία της απόσυρσης ε, της οδηγίας της άδεια μητρότητας δεν είναι μόνο κόλαφος εις βάρος των ε, ε, γυναικών και των ανδρών αλλά και κόλαφος εις βάρος της κοινωνικής Ευρώπης. Πώς θα εξηγήσετε στους πολίτες μας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει όταν μία από τις λίγες χειροπιαστές προτάσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη επί χρόνια αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και που απέτυχε και πάγωσε ε, εξαιτία τη τάση σα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχθούμε. Και η άγνοια όσον αφορά η παραμέληση των θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, όταν το Ευρωκοινοβούλιο έχει τεθεί υπέρ τη βελτίωση τη προστασία των γονεϊκών δικαιωμάτων, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε εδώ, πρόκειται και για τι μητέρε όμω και για του άνδρε, αναμένουμε το Συμβούλιο να αρθεί στο ύψος των υποχρεώσεών του και να ανταποκριθεί και με σοβαρό τρόπο να προβληματιστεί και να διαπραγματευτεί για τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη. Για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Γιούτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, γνωρίζουμε ότι ένα από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χαμηλή υπογεννητικότητα. Είναι ενισχυτικά τα δεδομένα σε όλα τα κράτη-μέλη. Η παλιά Ευρώπη ε, έχει ε, γενετικότητα σχετικά εντάξει μόνο χάρη στη μετανάστευση. Ωστόσο δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και μετά από χρόνια στασιμότητας πάμε να αποσύρουμε την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Εμείς ε, αντιτιθέμεθα σε αυτό το σκάνδαλο. Το Συμβούλιο ποτέ δεν συμπεριέλαβε στην ημερήσια διαταξή του το θέμα αυτό και η Λετωνική Προεδρία ούτε καν καταδέχτηκε να παρουσιάσει και να έρθει να μιλήσει στην Επιτροπή ΦΕΜ για το θέμα της έδειας μητρότητας που δεν είναι διακοπές. Ε, για αυτό το θέμα υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Καλό θα ήταν ίσως να μετριάσουμε λιγάκι τις προσδοκίες που προβλέπει το Κοινοβούλιο, αλλά να δώσουμε κάποιο αποτέλεσμα, ε, για να δώσουμε μια απάντηση στις, Ευρω... στις γυναίκες της Ευρώπης. Φτάνουν οι διακρίσεις που οι εργοδότες πολύ συχνά υποχρεούνται να κάνουν λόγω ελήψεως πολιτικών και φτάνουν οι διακρίσεις πια με τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες και μπορούν και οι γυναίκες που περνούν την περίοδο ε, της εγκυμοσύνης ε, ε ως ε, προθάλαμο της ανεργίας τους. Συμφωνήσαμε όλοι στις διάφορες συζητήσεις επ' ενός κειμένου το οποίο μας οδηγεί σε μια ίσως απόσυρση χωρίς νέα νομοθετική πρόταση. Να ζητήσω από την συγκεκριμένη την κυρία Ρένα και από τους συναδέλφους των άλλων ομάδων πώς γίνεται να απορρίπτουμε ένα ψήφισμα το οποίο απλά δίνει μια αιτιολογία στην Κομισιόν να αποσύρει την οδηγία. Γιατί δεν κάνετε μια νέα νομοθετική πρόταση όταν έχουμε ήδη μία στην οποία ε, μπορούμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση και την οποία θέλετε να εγκαταλείψετε προκαταβολικά. Εμείς θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες των πρασίνων αλλά να ρωτήσω τις άλλες ομάδες τι θα κάνετε. Για ποιο λόγο αλλάξατε πορεία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μάγερ, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί χρόνια υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για την άδεια μητρότητας. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πείσει τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν. Η συζήτηση για τις 18 ή τόσες εβδομάδες είναι μια συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί στα εθνικά κοινοβούλια και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου υπάρχει υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Α μην υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάμειξη. Ας έχουμε μια πιο δίκαια Ευρώπη, όπω υποσχέθηκε ο κ. Τίμερ μα. Μετά από τα λόγια, α ακολουθήσουν οι πράξει. Αναφέρθηκε η απόσυρση αυτή τη οδηγία. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να υιοθετούν τι δικέ του ρυθμίσει προ όφελο τη ανταπόκριση ε, προ τα συμφέροντα των ε, γυναικών και των ανδρών. Και η πρόταση προσευχή πρέπει να καταλήξει στην καλάθο των αχρήστων. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Έχει φτάσει επιτέλους η στιγμή να μιλήσουμε για κοινή γονική άδεια και όχι άδεια μητρότητας. Για να υποστηρίξουμε τις εργαζόμενες μητέρες πρέπει να εμπλέξουμε και τους πατέρες να, λάβουν, να αναλάβουν την ευθύνη ε, για τα μωρά τους και να μην υποχρεώνουμε τις γυναίκες να μείνουν στο σπίτι. Αυτό ακριβώς χαιρετίζω την... Ε, ε, ε, ε, την ανάκληση της οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο μητέρες στο σπίτι. Θα ήταν κατά τη γνώμη μου ένα μειονέκτημα και όχι μια πρόοδος. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες για να έχουν έναν ισορροπημένο βίο. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τις γυναίκες ως το μοναδικό γονιό που είναι υπεύθυνο για τα παιδιά και να ενθαρρύνουμε και δύο γονείς να αναλάβουν την ευθύνη των παιδιών τους. Το ε, και το πότε δεν πρέπει να λαμβάνεται ως απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είμαστε διαφορετικοί. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις οικογενειακές πολιτικές στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να έχουμε μία λύση που να ταιριάζει σε όλους 18 ε, ε, εβδομάδες υποχρεωτική άδεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι γυναίκες πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό όταν μπορούν και οι, οι, οι σύντροφοί τους να μείνουν σπίτι, όπως γίνονται στις βόρειες χώρες ημέρες. Ε, για παράδειγμα, αυτό ήταν ο λόγος που στη Σουηδία δεν ε, προωθήθηκε η άδεια μητρότητα, αλλά πατρότητα, ε, γιατί υπήρξε μία άποψη ότι η άδεια μητρότητα και η σχετική ρύθμιση ουσιαστικά παραβιάζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε στερεότυπα και σε σχέση με τη γονεϊκή άδεια. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκαρθία Πέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιοι συνάδελφοι σε αυτό το σώμα φαίνεται ότι δεν πληροφορήθηκαν για το τι πράγμα συζητούμε. Συζητούμε για νομική ρύθμιση που θα διασφαλίζει την προστασία της υγείας των γυναικών, μητέρων, εργαζομένων που θα είναι σύμβατη με την νομοθεσία εκείνη που θα προωθεί την συμφιλίωση της εργα... του εργασιακού βίου και του οικογενειακού βίου και θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της ε, ε, μητρότητας. Τοποθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλες τις μεγάλες μας διαφορές συμφωνήσαμε. Αυτή η συζήτηση είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στο η οδηγία αυτή να είναι πραγματικότητα και να μην τη συζητάμε πλέον ακόμα. Και απέχει πολύ το Κοινοβούλιο από τη θέση του Συμβουλίου. Ακούστηκε. Ποια είναι όμως θέση του Συμβουλίου. Αν δεν είναι σε θέση να μας αναφέρουν ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία υπερασπίζονται. Είναι απουσία σεβασμού για την προώθηση των πολιτικών υπέρ τη υγεία των γυναικών που εργάζονται και τη συμφιλίωση τη εργασιακή με την οικογενική ζωή. Κάνουμε λόγο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πέρες. Το λόγο έχει η κυρία Βυσνιεύσκα για ένα λεπτό. Ε, dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια δημογραφική κρίση στην Ευρώπη, κυρίως ε, στην Πολωνία. Και πρέπει να κάνουμε κάτι πραγματικά. Πρέπει να προστατέψουμε τις γυναίκες και τις οικογένειες. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την οικογενειακή πολιτική, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τις μητέρες. Και, μεταξύ... και η πρόταση για 20 εβδομάδες ε, θα μπορούσε να ήταν μια καλή ε, λύση. Όμως ε, όχι επειδή με αυτή τη ρύθμιση αυξάνεται η εργασιακή ζωή των γυναικών. Όχι. Είναι καλύτερη λύση επειδή είναι μια καλή λύση για τα άλλα προβλήματα. Την υπεργύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη, στην κοινωνία μας. Χωρίς μια σύνθετη, ολοκληρωμένη οικογενειακή πολιτική δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να προσφέρουμε λύσεις σε αυτά. Την κρίση δημοκρατίας δεν θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε. Θα πρέπει να επενδύσουμε στις οικογένειες και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μητέρες, τις γυναίκες που εργάζονται και θα πρέπει η κοινωνία να διαμορφωθεί με τρόπο που να είναι βιώσιμη ε, στο μέλλον. Και γι' αυτό η οδηγία προστασίας ε, της γονεϊκής άδειας ε, που τροχοπεδείται από το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αναφέρω ένα στοιχείο. Σε πέντε χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30% οι περιπτώσει παρενόχληση των γυναικών λόγω μητρότητα. Ε, Πολλέ χιλιάδε γυναίκε ε, έχουν υποχρεωθεί να παραιτηθούν ή έχουν απολυθεί σε σχέση με θέματα μητρότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή που το Συμβούλιο ουσιαστικά δεν έχει εκφράσει κάποια άποψη και η Κομισιόν προτίθεται να αποσύρει την πρότασή της. Θεωρώ ότι είναι ντροπή, όχι γιατί θεωρώ ότι οι γυναίκε ε, πρέπει να προστατεύονται πιο πολύ από άλλου ή ότι πρέπει να προστατεύουμε την οικογένεια περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να εγγυηθούμε το, δίκαιο αυτοδιάθε... το δικαίωμα αυτοδιάθεση των γυναικών στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα. Οι γυναίκε να μπορούν να αποφασίζουν μόνε τι επιλογέ του. Η επιλογή που μα προτείνεται σήμερα δεν είναι επιλογή ουσιαστικά θεωρούμε ότι μετά από την έγκριση από αυτήν εδώ την αίθουσα ενός κειμένου όπως αυτό που προτείνεται από τον κύριο Ταραμπέλα ε, είναι κάτι που δεν καλύπτει το χάσμα που υπάρχει αυτή την διακριτική μεταχείριση των γυναικών στην Ευρώπη. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Σεμπαστιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει πέντε στόχους για την αύξηση το 2020. Θα αναφέρω δύο. Ποσοστό απασχόλησης 75%. Πράγμα το οποίο σημαίνει να αυξηθεί και ο αριθμός των εργαζομένων γυναικών. Δεύτερο, να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων σε κοινωνικό αποκλεισμό, πράγμα το οποίο πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες που είναι τα κύρια θύματα αυτού του αποκλεισμού. Ερωτούμε τους, το, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι χωρίς μια οδηγία για την προστασία των γυναικών που είναι, γίνονται μητέρες. Είπε επανειλημμένα ο πρόεδρος Γιούγκερ ότι τερματίζεται τώρα η λιτότητα και πρέπει να εργαστούμε για τα δικαιώματα των πολιτών. Έχετε την ευκαιρία να αποδείξετε ότι πράγματι επιθυμείτε να το κάνετε αυτό. Η γονεϊκή άδεια, μητρική και πατρική, υπέρ όλων των οικογενειών στην Ευρώπη, υπέρ του έργου στο Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη μιας ελάχιστη συμφωνίας που δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε να υποβαθμίσουμε. Αν ε, ε αυτή την πρόταση, αν δεν τη δεχτείτε, εγκαταλείπετε τις γυναίκες και δεν τις βοηθάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι η υπογεννητικότητα. το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση στις χώρες εκείνες των οποίων η οικονομία δεν είναι σε καλή κατάσταση. στην ελλάδα η οποία υποφέρει από τους επώδυνους και επαχθείς όρους του μνημονίου για πρώτη φορά το 2013 ο αριθμός των θανάτων ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των γεννήσεων. ενώ λοιπόν στην ευρώπη η υπογεννητικότητα είναι γεγονός ενώ κατακλείζονται οι χώρες της ευρώπης από πλήθος παρανόμων μεταναστών με κίνδυνο στο άμεσο μέλλον να γίνουμε μειονότητα στη χώρα μας το συμβούλιο δεν εγκρίνει την επέκταση της αδείας μητρότητα στις είκοσι εβδομάδες διότι θα υπάρξει οικονομικό κόστος. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι αυτό είναι τραγικό όχι μόνο να το λέμε αλλά ακόμη και να το σκεπτόμαστε. η μητρότητα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το βλέπουμε με την δέουσα προσοχή και σοβαρότητα δεν έχουμε το δικαίωμα τόσο απέναντι στο έθνος όσο και απέναντι στο κράτος να αρνηθούμε την συνέχεια της ζωής του στο μέλλον. πρέπει να στηρίξουμε πάση θυσία τη, μικρότητα, τη μητρότητα. δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε στους απογόνους μας είτε να δουν το φως της ζωής είτε εάν γεννηθούν να μην μπορούν να ζήσουν ως ελεύθεροι και πολιτισμένοι άνθρωποι. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Χιμένεφ Μπεφερίλ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία έχει ως στόχο να εφαρμοστούν μέτρα για να βελτιωθεί η υγεία στην εργασία των εγγύων εργαζομένων, εκείνων που έχουν γεννήσει και εκείνων που θυλάζουν. Είναι μια οδηγία για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία. Δεν κατανοώ για αυτούς τους λόγους τη σιωπή του Συμβουλίου και που δεν είναι δυνατόν οι γυναίκες να εγκαταλείψουν το δικαίωμα του να έχουν παιδιά και να εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας τους δεν μπορεί να είναι εμπόδιο τα παιδιά στο να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή απασχόληση οι γυναίκες. Ξέρω δεν είναι εύκολο να προχωρήσει κανείς ε, σε έναν κόσμο όπου αλλάζουν και διαφέρουν τα πράγματα σε σχέση με τις διατάξεις για τα εργασιακά θέματα από χώρα σε χώρα. Όμως το Ευρωκοινοβούλιο τοποθετήθηκε με σαφήνεια και είπε ότι πρέπει να επανεξεταστούν οι εργασιακοί όροι και συνθήκες απασχόλησης των εγγύων γυναικών. Η συμφιλίωση ε, της ε, εργασιακής ζωής και της οικογενειακής ζωής σημαίνει να βοηθήσουμε στο να προοδεύσει η Ευρώπη όταν θα έρχεται η ώρα να επιμερίσουμε το έργο και τις ευθύνες μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και ανασφάλειας όσον αφορά το εργασιακό μέλλον σε σχέση με τη γέννηση ενός παιδιού και θα πρέπει να ασκηθεί πίεση ώστε να αλλάξει η θέση και η στάση που υιοθετείται σήμερα από το Συμβούλιο και για κάτι το οποίο ε, το Κοινοβούλιο Συμβούλιο έχει υιοθετήσει πρέπει να αναζητηθούν οι καλύτερες λύσεις γι' αυτό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Χέντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα τη μη διακριτική μεταχείριση είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την εγκυμοσύνη και την αδημητρότητα. Έχει μεγάλη ιστορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1985 με μια συμφωνία που αφορούσε τη μη διακριτική μεταχείριση βάσει τη ε, εγκυμοσύνη και τη αδεσμητρότητα. Παρά αυτή την αρχή τη μη διακριτική μεταχείριση, αντιλαμβανόμαστε ότι οι γυναίκε ακόμα σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, ειδικότερα στο χώρο εργασία. Το βλέπουμε κυρίως ε, στο θέμα των συζητήσεων για την αδημητρότητα και εδώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα. Μπορούμε να παρουσιάσουμε νούμερα 60%, 30% ανάλογα με την ε, κατάσταση. Ε, η πλειοψηφία των γυναικών έχει να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και πολλές ανησυχίες όσον αφορά το γύρας. Επίσης πολλές γυναίκες ε, δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα στις ε, προσωρινές θέσεις εργασίας ε, δυσκολεύονται οι γυναίκες να αμυθούν κατά διάρκεια της εποχής όπου πρέπει να προσέχουν τα παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω αδιασμητρότητας ή εγκυμοσύνης. Για μένα είναι θέμα αλληλεγγύης με τα... γυναίκες τη Ευρώπη. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση βλέποντα πραγματικέ συνθήκε στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, η κυρία Ζητνάνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση για την παράταση της άδειας μητρότητας ουσιαστικά ήθελε να δημιουργήσει μια καλύτερη κατάσταση για τις μητέρες, εργαζόμενες μητέρες, ώστε να βοηθηθούν στην εργασιακή αγορά να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Μετά όμως από 7 χρόνια δεν υπάρχει όμως κάποιο συμβιβασμός που να είναι δεκτός από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από ε, την αρχή πάλι, από μηδενικού σημείου. Όμως, η ε, δυνατότητα να είναι αποδοτικές οι ευρωπαϊκές οικογένειες ε, δεν εξαρτάται μόνο από την γονεϊκή άδεια. Χρειάζονται επίσης και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς θέσεις για τα παιδιά τους οι γυναίκες και κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις. Το αν θα δημιουργηθεί ή όχι αυτή η κατάσταση εξαρτάται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα για την ανευθυνότητα και την ενοχή του αυτέξιμου Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Ωστόσο, θέλω να επικεντρωθώ στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπω είπε η Επίτροπο, πράγματι έχει τον στόχο να αποσύρει αυτή την πρόταση. Αν αποσύρεται αυτή την πρόταση οδηγία, θα καταλήξετε σε δύο σημαντικότατα σφάλματα. πρώτον, σε σχέση με την υπέρβαση, την αγνώση των δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Και μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θέλει να προαγάγει την κοινωνική Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Σε σχέση με τον θεματοφύλακα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Το δεύτερο, δεύτερο σφάλμα δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό προηγούμενο διότι δεν θα είναι δυνατόν να υπάρξει η έγκριση από το Συμβούλιο όταν δεν υπάρχει έγκριση αποσύρετε εσείς μια πρόταση. Πολύ σημαντικό σφάλμα. Με τη δική μας υποστήριξη πρέπει να συνεχίσετε να πιέζετε το Συμβούλιο για να προαχθεί αυτή η οδηγία. Με την απόσυρση της οδηγίας τι γίνεται. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε χρήση αυτού του, αυτής της δυνατότητας εσείς. Είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Σούιτσα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 Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα το Συμβούλιο θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Πέρασαν τόσα πολλά χρόνια μετά από την πρώτη οδηγία και συνένεση δεν επετεύχθη. Όμως επίσης ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου όταν ζητεί μια νέα κίνηση τι νέο θα μπορούσε να συνεισφέρει μια νέα ε, κίνηση σε σχέση με αυτή την οδηγία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο που να μπορεί να προσθεθεί χωρίς να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας. Όμως γνωρίζουμε ότι η κοινωνική πολιτική και η οικογενειακή πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση εκάστοτε των κρατών μελών. Ποια είναι εκείνη και πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη αυτά τα θέματα. Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία βλέποντας ιδιαίτερα σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα το τι συμβαίνει για την Κροατία πρέπει να πω ότι έχουν 26 εβδομάδες ε, άδεια μητρότητας οι γυναίκες, οι εργαζόμενες γυναίκες και με τους επόμενους έξι μήνες ε, με χαμηλότερες απόλαβες. Και οι άνδρες, ε, οι σύζυγοι μπορούν να αποφασίσουν αν και εκείνοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος πατρότητας ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να επωφεληθούν. Για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει με σαφήνεια να εκφράσουν την άποψή τους στο Συμβούλιο και να δοθεί συνέχεια. Και αν δεν είναι σε θέση να το πράξουν αυτό, ε, τότε τουλάχιστον να υπάρξει μια νέα οδηγία, η οποία θα υποστηρίζει όμως τις θέσεις των κρατών μελών. Λυπούμε που υπήρξε μια διακοπή, διότι αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο ε, ε, διέκοψε τη συνέχεια της σκέψης. Τη δέχεστε. Σα ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε την μπλε κάρτα μου. Αναφέρατε την Κροατία και χαίρομαι που την αναφέρατε. Διότι ήθελα εγώ να κάνω λόγο για την κατάσταση ε, στην Κροατία. Έχουμε καλά παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία είναι ένα από αυτά τα καλά παραδείγματα. Σα ερωτώ λοιπόν, συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι απίστευτο ότι κάτι, κάποια πλουσιότε, πολύ πλουσιότερα κράτη-μέλη από την Κροατία τροχοπεδούν την επίτευξη προόδου για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί αυτή την ε, ώρα που έχει προχωρήσει πάρα πολύ και που τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ συνάδελφε Γιάκοψη για την ερώτηση. Στοχεύει και στην ίδια κατεύθυνση προς αυτά που έλεγα πιο πριν για την οικονομική ενίσχυση της ε, ε, κοινωνίας που πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών και η Κροατία είναι ένα καλό παράδειγμα ως προς αυτά. Το Συμβούλιο θα πρέπει να προβληματιστεί για αυτό το θέμα, για αυτή την πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να ξεκινήσει απαρχήσα ε, από μια νέα αρχή αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να δοθεί συνέχεια στις διαβουλεύσεις. Οι γυναίκες έχουν δικαιώματα για ισότητα στους χώρους εργασίας τους πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να υπάρξει επίτευξη συνένεση για μια λύση που θα δίνει και θα διασφαλίζει αυτή την ισότητα για τις γυναίκες σε μια ελεύθερη ευρωπαϊκή κοινότητα. Η κυρία Thank you, Chair. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της συμπεριφοράς του Συμβουλίου που ήταν πραγματικά ε, πάρα πολύ κακή. Εδώ και πέντε χρόνια, όπως είπαν και προλαλήσατε συνάδελφοι, από τότε που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η οδηγία όλοι και η ομάδα μου, αλλά και η, όλη η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, το εγκρίναμε αυτό και το Συμβούλιο απλώς το μπλόκαρε, το αγνόησε, μια μικρή μειοψηφία μπλόκαρε την οδηγία και πρέπει να αναρωτηθεί κανείς γιατί, γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, για ποιο λόγο υπήρξαν αρκετά κράτη-μέλη που το καθυστέρησαν για πέντε χρόνια και το μόνο συμπέρασμα λογικό που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου Κοινοβουλίου κράτη-μέλη που δεν θέλουν την ομοθεσία αυτή, που δεν θέλουν την ισότητα των φύλων και δεν θέλουν ε, να υπάρχει προστασία των αγγείων γυναικών στο χώρο εργασίας. Δεν είναι μόνο απαράδεκτος άποψη, είναι και πάρα πολύ κοντόφθαλμο γιατί αυτή η οδηγία θα έδινε τη δυνατότητα στι στις γυναίκες ε, να μπουν στην αγορά εργασίας ε, με πολύ καλύτερη οικονομική επίδοση και αυτό θα ήταν πολύ επικερδές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα λεπτό η κυρία Φων Στόρχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνουμε σήμερα λόγο για την άδεια μητρότητα και πώ μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν συμμετείχε το Συμβούλιο, πράγμα που δεν συμβαίνει και δεν συμμετέχει. Είναι καλό και αυτονόητο οι γυναίκες να προστατεύονται όταν εργάζονται. Φυσικά πρέπει να προστατεύονται Ωστόσο όμως απορρίπτω την τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δύο λόγους. Πρώτον, η οδηγία στην μέλουσα μητέρα βλέπει πάντα μια εργαζόμενη. Την εγκυμοσύνη την θεωρεί ω πρόβλημα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον χώρο εργασίας. Αυτό είναι μια πολύ μαρξιστική προσέγγιση η μητρότητα ως ελάττωμα για την αποδοτικότητα εργασίας της γυναίκας. Δεν είναι όμως η μητρότητα βάρος για την κοινωνία. Μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά, για την κοινωνία, για τις οικογένειες και στο τέλος τέλος για την, για την οικονομία. Η μητρότητα λοιπόν είναι εκείνη που οδηγεί στο να προαφεί η οικονομία και να καταστεί ισχυρή. Δεν είναι λοιπόν όμως αρμόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μητρότητα. Μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμίσουν τα σχετικά θέματα. Ελπίζω να μπορούν να το καταφέρουν όμως αυτό. Το λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Κόμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Μιλάμε για την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών στη χώρα εργασία σε κρίσιμε εποχές ε, σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους όταν δημιουργούν ζωή. Δεύτερον, έχουμε το σημερινό πλαίσιο με την υπογεννητικότητα που μεγαλώνει όλο και περισσότερο, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Με όλα αυτά, ο Ευρωπαίος νομοθέτης έπρεπε να νομοθετήσει γρήγορα. Αντί γι' αυτό όμως έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεων λόγω του Συμβουλίου. Υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα και πρέπει να βρούμε κάποια ισορροπία. Πρέπει να υιοθετήσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σεβόμενη την επικουρικότητα και τις διάφορες εθνικές παραδόσεις. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε μια ακινησία χωρίς προοπτική. Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι λόγω προσωπικών συμφερόντων χωρίς να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. Κυρία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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Ρένα, την εισηγήτριά μα, για την επιμονή που έδειξε σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώ δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ω προ τη σημασία που έχει για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ κατεπήγον αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για το θέμα αυτό, για να μην υπάρχουν πια διακρίσει. Για ποιο λόγο το Συμβούλιο έκανε τόσα λίγο, γιατί δεν υπήρξε επικοδομητικό διάλογο, γιατί τονική Προεδρία δεν άκουσε τα αιτήματα των κρατών μελών για τη συζήτηση αυτών των, ε, θεμάτων. Θα έπρεπε να λάβει, να λάβει θέση το Συμβούλιο και όχι να κοφεύει. Ε, όσον αφορά τώρα ε, που μας ε, δημιουργεί πρόβλημα το θέμα του κόστους δεν έχουμε ποτέ πει ποιο είναι το κόστος της μη δράσης ειδικότερα όταν πρόκειται για την άδεια της μητρότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό κείμενο το οποίο προστατεύει τις γυναίκες στο χώρο εργασίας ε, και συμπεριλαμβάνω και σε αυτό τη διάσταση της μητρότητας. Ε, έχει άμεση σχέση με το θέμα της κοινωνικής προστασίας, της ισότητας των πολιτών ναι, αλλά συγγνώμη, το 2008 γνωρίζαμε όταν έγινε η ψηφοφορία σε επίπεδο κοινοβουλίου ότι μπαίναμε σε ένα πάρα πολύ ολισθηρό έδαφος. Η δική μας ευθύνη είναι να παραμείνουμε δεσμευμένοι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή τι θέλουμε να επιτύχουμε. Σήμερα δεν άκουσα ούτε ομοφωνία ούτε σύγκληση για, το, για το, τη βούλησή μας. Πρέπει νομίζω να γυρίσουμε σελίδα, να ξαναρχίσουμε με στέρεα βάση, γιατί δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι άκουσα σήμερα τίποτε που να μας, μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε μια πραγματική, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις γυναίκες. Ναι, έχουν πολύ καλή εκπαίδευση γυναίκες, ναι, έχουν δικαίωμα ε, στην εργασία, ναι, ήταν θύματα της κρίσης και πρέπει μέσα μέσα, από ένα νέο κείμενο να τις βγάλουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Στάιρουκ. Για να εξυγχρονίσουμε την οικογενειακή πολιτική και να ενθαρρύνουμε το ρόλο του πατέρα στη διαδικασία είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά εδώ μιλάμε για την προστασία της υγείας ε, και της εργασία. Δεν αφορά το θέμα μόνο να προστατεύουμε τις μητέρες και τα παιδιά πριν και μετά τη γέννα. Το ζήτημα αυτό αφορά τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Το να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα παίζουν ε, πλήρη ρόλο στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα πρόσφατο κομμάτι όλο αυτού. Τα ελάχιστα πρότυπα που ε, εφαρμόζει ο ILO πρέπει να εφαρμόζονται και στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε ε, ένα κοινό ενισχυμένο σύστημα προστασίας για τις μητέρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θα στείλει ένα χειρό και σωστό μήνυμα για να σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε θέματα κοινωνικής ε, δικαιοσύνης. Για ένα λεπτό η κυρία Κομοντίνη Κατσία. Grazie, Sir President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει αυτή την οδηγία πολλές φορές ε, ε, αντικατοπτρίζει τις κοινωνικο-οικονομικές πραγματικότητες στα κράτη-μέλη και στην Ένωση. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτή την οδηγία χωρίς να θυμόμαστε τα εξή. Τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει γύρανση του ε, πληθυσμού και υπογεννητικότητα. Ορισμένα κράτη-μέλη δυσκολεύονται να προσελκύσουν τις γυναίκες στην αγορά εργασίας ή να τις βοηθήσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους όταν φτάνουν σε ηλικία τεκνοποίησης. Εμείς τονίζουμε διαρκώς ότι οι γυναίκες είναι ίσα μέλη στον κόσμο. Είμαστε υπέρ της ισότητας των φύλων. Ζητάμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τις εργαζόμενες μαζί με το δικαίωμα συμφιλίωσης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και μετά δεν καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε επί πολιτικών που ε, αφορούν αυτές τις κοινωνικο-οικονομικές πραγματικότητες. Η πρόταση της Κομισιόν για απόσυρση αυτού του φακέλου δεν ικανοποιεί πολλούς, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του αδιεξόδου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αρχές που ανέφερα όμως μέσα σε όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε άλλα μέτρα για να τα οποία θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε. Ένα λεπτό η κυρία Γιουγκέριος. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι ότι οι πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση ενός παιδιού είναι κρίσιμες εβδομάδες. Κατά τις εβδομάδες αυτές βλέπουμε κατά πόσο ο πατέρας θα βοηθήσει στον οικοκυριό και αν η μητέρα μπορεί να εργαστεί ε, πλήρως. Και αυτό χρειαζόμαστε ένα πολύ καλά ρυθμισμένο πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη ζωή του παιδιού και της μητέρας και του πατέρα. Και είναι μια αποφασιστική πτυχή για την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Και είναι απογοητευτικό να βλέπει κανείς ότι για το Συμβούλιο οι έγκυες γυναίκες είναι απλώς σε ένα παράγοντα κόστους ε, και ότι το καλύτερο είναι να αποσυρθεί αυτή η πρόταση χωρίς να ληφθεί υπόψη η δήλωση του ε, δικαστηρίου. Εμείς δείξαμε ότι θελήσαμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση και γι' αυτό ακριβώς ζητούμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσεγγίσουν τη δική μας θέση. Η ε, μονομερής ε, ανάκληση σίγουρα δεν είναι ε, μια καλή εξέλιξη. Πρέπει να δοθεί μια πραγματική δυνατότητα στις γυναίκες να καλύψουν την καθυστέρησή τους. Ευχαριστώ. Μια Ευρώπη που θέλει να αναπτυχθεί πραγματικά θα είναι μια Ευρώπη που θα υποστήριξει μια ιδέα ανάπτυξη που θα μπορεί να προωθήσει δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ίση πρόσβαση και ίσε ευκαιρίε. Με την αξιοποίηση του, κεφαλαίου των γυναικών σημαίνει δημιουργία πολιτικών συμφιλίωσης και, κοινής... Ε, και κοινού επιμερισμού των ευθυνών. Γι' αυτό οι έδειε μητρότητα και πατρότητας ε, αποτελούν όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. Μέσω του νέα φιλοσοφίας εργασία, υψηλή ποιότητα που δεν αποκλείει κανέναν ε, στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας την πρόθεση μια δίκαιη Ευρώπη γυναίκε. Απαράδεκτη η στάση όσον αφορά την αδιαμητρότητα από το Συμβούλιο διότι τα κίνητρα είναι θεωρώ εγώ υποκριτικά. Γι' αυτό ε, υποστηρίζω τη συνέχιση του διαλόγου ο οποίος θα πρέπει να συνεχιστεί γρήγορα και να γίνει σωστά. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί δέκα αιτήματα. Προτείνω να αφαιρεθούν οι συνάδελφοι που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα της ερώτησης μέσω της μπλε κάρτας, οπότε μένουμε στους 7. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν και οι 7, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί αυστηρά από όλους ο χρόνος του ενός λεπτού. Προχωρούμε με την κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι όλους ιδιαίτερος ε, που η χώρα μου είναι η Τσεχία, όπου 28 εβδομάδες είναι η άδεια μητρότητας και οι γυναίκες λαμβάνουν 70% του μισθού τους κατά τις εβδομάδες αυτές. Ξέρω όμως ότι η κατάσταση διαφέρει στα άλλα κρατημέλη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε ελάχιστες ε, προδιαγραφές ε, στον, ε, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας να υπάρχει ε, σωστή φροντίδα των εγγύων γυναικών και των οικογένειών τους. Είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης, είναι η επένδυσή μας για το μέλλον και Ελπίζω ότι η περαιτέρω δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποστηρίξει τις ε, εργαζόμενες γυναίκες και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους της. Ευχαριστώ. Μιλάμε συνεχώς για ισότητα δικαιώματα, ισότητα φύλων, δικαιώματα αναπαραγωγή, αλλά το πολιτικό βάρο αυτού του θεσμικού οργάνου δεν φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό για να βοηθήσει να συμφιλειώσουν οι γυναίκε στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Αρένα για την αιμονή ε, ε, τη και την αποφασιστικότητά τη. Όπω φαίνεται στην Ευρώπη δεν συμφωνούν όλοι στο να φροντίσουμε να υπάρχει αμοιβόμενη ε, ε, άδεια μητρότητα πριν και μετά τη γέννηση. Μα τι άλλο να ζητήσουμε από τι γυναίκες, να περιμένουμε οι αρχηγοί ε, κρατών και κυβερνήσεων, κυρίω άνδρε, να χορηγήσουν αυτή τέτοιο δικαίωμα στι γυναίκε το να είναι μητέρα κάποια γυναίκα δεν είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα. Είναι απαράδεκτη η στασιμότητα αυτή για την οδηγία αυτή περί της μητρότητας. Δείχνει ότι υπάρχει τεράστια πολιτική ε, έλλειψη βούλησης ε, για τις γυναίκες. Ο πρόεδρος Γιουνκέρ ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει η Κομισιόν μια νέα πρωτοβουλία πιο συγχρονή και δεν γνωρίζουμε τους όρους και τις διατάξεις της και στο μεταξύ οι δυσκολίες των γυναικών δεν πάβουν να υπάρχουν όπως ανέκαθεν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η διγλωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσεύει. Η Τρόικα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της Κομισιόν κατά τη διάρκεια του μνημονίου επέβαλε μείωση των μισθών, κατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Τώρα επειδή το Συμβούλιο διαφωνεί, η Κομισιόν με τον κύριο Τίμερμανς αποσύρει την νομοθετική ρύθμιση για την εναρμόνιση της άδεια μητρότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι στο όνομα της δίθεν βελτίωσης της νομοθεσίας η Κομισιόν πετά την άδεια μητρότητα στον κάλαθο των αχρήστων όμως οι γυναίκες όπως και οι νέοι είναι τα μεγάλα θύματα της κρίσης. χωρίς προστασία των γυναικών που γίνονται μητέρες δεν μπορεί να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες των γυναικών στην εργασία. ταυτόχρονα η απόσυρση της οδηγίας θα εντείνει την κρίση υπογεννητικότητας στην ευρώπη και κυρίως στις χώρες του μνημονίου στη φτωχοποιημένη από το μνημόνιο ελλάδα το 2013 μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 6,21%. είκοσι ένα ενώ σύμφωνα με έκθεση των γιατρών του κόσμου στην ελλάδα τέσσερι στις δέκα γυναίκες θα γεννήσουν ένα παιδί λιγότερο από ό,τι προγραμμάτιζαν. ταυτόχρονα η τρόικα με την πολιτική της θεωρεί τα παιδιά τεκμήριο που αυξάνουν το φορολογικό βάρος της οικογένειας. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Συμβούλιο πρέπει να αποτροχοπεδίσει την οδηγία για την άδεια μητρότητας και πρέπει να προβληματιστεί για αυτό το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση Κατανοούμε αυτό το θέμα, αλλά αυτό και άλλα θέματα πρέπει να δώσει κίνητρο να υιοθετηθεί μια άλλη στάση και τοποθέτηση αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναχρονισμός να συνεχίσει ως λέσχη φίλων το Συμβούλιο, θέλοντας να διατηρήσουν κάποιες δομές εξουσίας που έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα και πρέπει να αφουγκραστούν τους πολίτες για την επίλυση των προβλημάτων. πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα γυναικών ή μητέρων. Χρειάζεται αυτή η πρόταση για να αντιμετωπιστεί η δημογραφική συρρήκνωση. Αν δεν γίνει αυτό, παραβιάζουμε θεμελιώδη δικαιώματα. Μειώνεται και υποβαθμίζεται η ανταγωνιστικότητά μα. Και τέλο τέλο διακυβεύεται το καλύτερο μέλλον που επιθυμούμε για όλου. Διερωτήθηκε το Συμβούλιο πόσο στοιχίζει η ανισότητα που είναι το μόνο που μα προτείνουν. Και όταν λένε ότι είναι διαφορετικέ οι προοπτικέ και οι προσδοκίε. Ποιε είναι οι προσδοκίε του Συμβουλίου, ήθελα να το μάθω. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ζαριανόπουλος. Η συνολική ευρωνοσιακή πολιτική για τη γυναική εργασία και η απόρριψη της οδηγίας για την άδεια μητρότητας από κυβερνήσεις και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύουν τη βαρβαρότητά τους, καθώς θυσιάζουν ακόμα και αυτήν για τη μείωση του εργατικού κόστους. Αυτή είναι η λεγόμενη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής έτσι ενισχύεται η εργοδοτική τρομοκρατία με απολύσεις γυναικών λόγω μητρότητας πριν από αυτήν κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. όλα αυτά θα σημάνουν πισωγύρισμα ακόμα και σε κράτη μέλη που ισχύει μεγαλύτερη άδεια όπως για παράδειγμα στην ελλάδα καταργήθηκε ήδη το επίδομα τοκετού. οι εργαζόμενες γυναίκες στα νέα ζευγάρια δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από διαπραγματεύσεις και υποσχέσεις. τώρα οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρα για ουσιαστική προστασία της μητρότητας της υγείας των γυναικών στους χώρους δουλειάς σταθερή δουλειά με δικαιώματα αποκατάσταση επιδομάτων απαγόρευση απολύσεων και άδειες μητρότητας ανάλογες με τις ανάγκες της μητέρας και του παιδιού αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τη λαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Νέκοφ. Уважаеми господин председател, въпреки Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πολλές εκκλήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο όπου λέμε ότι πρέπει να επανεδιαπραγματευτούμε αυτή την οδηγία και όπως βλέπουμε δεν έχει επιτευχθεί τίποτα. Έχει έρθει η ώρα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες στην Ευρώπη, όσες γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν παιδί. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια, να επιτύχει κάποια ισορροπία μεταξύ συνομοθετών. Δεν είναι περίεργο που η νομοθεσία στον τομέα αυτό έχει μείνει απαράλλακτη τα τελευταία 20 χρόνια. δεν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για καλύτερα επίπεδα, για καλύτερη διοικητική διαχείριση, διότι το διακύβευμα εδώ δεν είναι μόνο η υγεία των γυναικών. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σημαντικά δημογραφικά προβλήματα. Θα χρειαστεί να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να κάνουν παιδιά και πρέπει οπωσδήποτε να εθετήσουμε αυτήν την οδηγία. Παρακαλώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αρένα. Αξιότιμοι συνάδελφοι, όλες οι παρεμβάσεις εκτός από εκείνη από την Τσεχία ήταν και είναι κόλαφος κάθε γυναίκας και των πατέρων μια θρασίτητα τι συμβαίνει σε βρεφονιπιακούς σταθμούς πληρώνουν ε, οι άνθρωποι για αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι δωρεάν. Τι σημαίνει άδεια μητρότητας. Δεν είναι άδεια. Θα έπρεπε να πληρώνεται. Να έχει parental wages, δηλαδή μητρικό μισθό. Αυτό θα ήταν μια ε, σωστή κίνηση. Μια νέα κίνηση τώρα. Επιτροπή και Συμβούλιο. Έχετε το θάρρος για μια νέα κίνηση. Ο χρόνος της γονεϊκής άδειας δεν είναι άδεια. Είναι περίοδος μισθού. Είμαστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής οικογενειακής στρατηγικής οι εργοδότες θα πρέπει να μην θεωρούν την άδεια μητρότητας ως απώλεια μητρότητας και πρέπει εδώ να δούμε και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι όταν πληρώνεται μισθός για τους γονείς αυτό είναι θέμα απασχόλησης και ανήκει στα κοινωνικά θέματα και στα θέματα απασχόλησης. Οι γυναίκες, οι μητέρες μέσα στο δημογραφικό πλαίσιο είναι οι πιο δυνατοί, ισχυροί παράγοντες δυναμικού. Ευχαριστώ. Ε, έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. πριν περάσουμε στο κλείσιμο της συζήτησης. Να μας πείτε μήπως αλλάξατε και γνώμη μετά πώς ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. αποτέλεσε πηγή έμπνευση για μένα αλλά και πηγή ενθάρρυνση. Σκεφτόμουν ε, τα όσα λέγατε και είπατε ότι μιλάμε εδώ για την ε, νομοθεσία για τα δικαιώματα των γυναικών. Και η ερώτησή μου είναι το να κάνει κανείς παιδιά είναι χόμπι ή πολυτέλεια που οι γυναίκες μπορεί να, μπορούν να έχουν ή όχι. Ε, ή μήπως θα χρειάζεται τα παιδιά η κοινωνία. Πώς είναι δυνατόν οι γυναίκες να αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο της ζωής τους στο να εργάζονται δωρεάν, ουσιαστικά φροντίζοντας τα παιδιά. Είναι μια δουλειά που χρειάζονται αυτές ή μια δουλειά που χρειάζεται η κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι ότι για αυτή, για αυτή την αρχή στην οποία αναφέρθηκα και για την οποία δεσμεύτηκα ε, πρέπει να βρούμε ένα νέο παράδειγμα. Πρέπει να το να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό μόνο από την άποψη των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν αρκεί. Όταν μιλάω για προώθηση της πολιτικής ισότητας των φύλων, αντιλαμβάνομαι ότι τα επιχειρήματα που αναφέρονται σε ισότητα, μη διακριτική μεταχείριση των γυναικών, είναι επιχειρήματα τα οποία είναι ζητήματα που αφορούν ε, καθαρά τη του φύλου είναι κάτι που αιτιολογεί τη στασιμότητα στην οδηγία αυτή για την αδιαμετρότητα. Γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει επικαιροποιηθεί αυτή η οδηγία τόσα χρόνια. Το πρόβλημα που έχει αυτή η απόφαση, το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην πρόταση απόσυρση της οδηγίας είναι ε, η διάρκεια, ο χρόνο που έχει διαρκήσει. Όπως είπα, πρέπει να δούμε επιχειρήματα και οικονομικά, όχι μόνο ισότητα των φίλων. Είναι φιλοσοφικό το ζήτημα. Εγώ είμαι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσω τέτοια επιχειρήματα οικονομικά. Κάποιο είπε ότι είναι μαρξιστικά τα επιχειρήματα αυτά. Δεν νομίζω. Κατ' εμέ, ένα καλό επιχείρημα θα ήταν να πούμε ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν να γεννούν φορολογούμενους. Ε, δεν είναι πολύ ωραίο βέβαια να το λέμε έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει νόημα. Αυτός είναι ο στόχος όταν έχουμε επιχειρήματα και θέλουμε να έχουν αποτέλεσμα. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι οι γυναίκες όταν δεν συμμετέχουν στην οικονομία επαρκώς και δεν κάνουν παιδιά, αυτό δημιουργεί πλήτη την οικονομία. Η κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα αποτελεί τροχοπέδι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά επιχειρήματα και τα οικονομικά. Υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι τα επιχειρήματα ε, περισσότερα των φύλων και μη διακριτική μεταχείριση των γυναικών πρέπει να είναι τα ισχυρότερα. Τώρα α δούμε την οδηγία ω έχει. Έχουμε δύο δυνατότητε για το μέλλον. Μπορούμε είτε να ε, σπρώξουμε αυτή την οδηγία που έχουμε το 2008 όπως είπε η κυρία Αρένα, ε, η οδηγία αυτή τουλάχιστον επιλέει κάτι πριν προκύψει κάτι νέο. Συμφωνώ με αυτό. Θα μπορούσαμε να επικυρωποιήσουμε αυτή την οδηγία ώστε να έχουμε τουλάχιστον κάτι, κάτι το οποίο να διασφαλίσει καλύτερη προστασία των μητερών και των γυναικών και σε τελική ανάλυση μπορεί να διασφαλίσει και καλύτερη αναγνώριση των γυναικών σε επίπεδο κοινωνία. Ίσως να ζητάμε πολλά εδώ από μια οδηγία, αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα ως επιτρόπου ω Επίτροπο. Ε, κατά την άποψή μου θα ήταν απλούστερο να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κρατη με εκείνα, που είναι πολύ άριθμα, ε, μεγάλη πλειοψηφία, ε, που αντιτίθεται να αλλάξουν θέση. Εγώ έχω κάνει την προσπάθεια. Προσπάθησα η οδηγία αυτή να φτάσει σε κάποια διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο ώστε να ξεμπλοκάρει. Όχι γιατί αυτό είναι ευκολότερο για μένα, αλλά γιατί συμφωνώ με την κυρία Ρένα και του άλλου συναδέλφου που θέλουν, αν μη τι άλλο, κάτι, έστω και λίγο. Η δεύτερη ε, δυνατότητα είναι η εξή. Το να παρουσιάσουμε κάτι καινούριο. Πριν μιλήσουμε για κάτι καινούριο, για το οποίο πολλοί λένε δεν ξέρουμε τι θα είναι, να σα πω τα εξή. Πριν ε, πάω στην Κομισιόν ζήτησα ανάλυση των επιπτώσεων τη οδηγία ε, περί άδεια μητρότητας στην απασχολησιμότητα και αντιληφθήκα ότι η νομοθεσία έτσι όπως έχει δεν επηρεάζει πραγματικά την απασχολησιμότητα. Αυτή η διαπίστωση είναι μάλλον οικονομική. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι από το 2008 πολλά κράτη-μέλη ενέκριναν νομοθεσίες που διασφαλίζουν καλύτερη προστασία των γυναικών. Και αυτό αποτέλεσε ε, αιτία για τη συμπεριφορά ορισμένων εκπροσώπων του Συμβουλίου, παρότι εγώ δεν μιλάω εκ μέρου του Συμβουλίου τώρα. Τώρα, αυτό το νέο τι μπορεί να είναι. Είναι ένα πολύ περίπλοκο τομέα αυτό. Εγώ είμαι φιλόδοξη. Και γι' αυτό το λόγο λέμε να αποσύρουμε αυτή την οδηγία για να παρουσιάσουμε κάτι πιο ε, αποτελεσματικό, κάτι πιο φιλόδοξο ε, σε δύο μέτωπα. Αφενός να διασφαλίσουμε τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Όχι μόνο κατά την περίοδο της μητρότητα, αλλά για όλη τη διάρκεια ζωής. Ε, στο πλαίσιο κάποιας αρρωγής προς τις οικογένειες ε, θέλουμε να μπλέκονται και οι άνδρες ώστε οι άνδρες να μπορούν να έχουν και αυτοί αυτή την πολυτέλεια. Ε, την πολυτέλεια του να παραμείνουν στο σπίτι και να φροντίσουν και αυτή την οικογένεια, αυτή την πολυτέλεια εντό εισαγωγικών που αυτή τη στιγμή δίνουμε μόνο στις γυναίκες. Και αυτό δημιουργεί ένα όλο και μεγαλύτερο οικονομικό χάσμα και αυξάνει την φτώχεια των γυναικών στην Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα πραγματικά περίπλοκο. Αυτή η συμφωλίωση τη οικογενειακή και τη επαγγελματική ζωή με συνέπειε όχι μόνο στη μη διακριτική μεταχείριση, αφορά και το ζήτημα τη εργασία, του δικαιώματο στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων υπάρχουν πολλέ και διάφορε θέσει στα διάφορα κράτη-μέλη λόγω της διαφορετικής θέσης των γυναικών σε κάθε κράτος, των διαφορετικών παραδόσεων. Σε άλλες χώρες οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο από τις άλλες. Στη δική μου χώρα συνήθως λένε ότι η γυναίκα αν αφού κάνει παιδί ε, γυρίσει γρήγορα στη δουλειά της δεν είναι καλή μητέρα. Σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι ακριβώς το αντίθετο. Να θυμηθείτε λοιπόν ότι ε, βρισκόμαστε σε πολυάριθμες, πολύ διαφορετικές καταστάσεις ε, σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Πρέπει να αναλύσουμε επίσης και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είπε κάποιος σε αυτήν εδώ την πλευρά της αίθουσας, πρόκειται και για αρμοδιότητες ε, κοινέ ε, σε ορισμένες ε, περιπτώσεις με τα κράτη-μέλη. Μία περίπτωση δεν θέλουμε να πλήξουμε την αρχή της επικουρικότητας. Κάποιο με ρώτησε πότε θα παρουσιαστεί αυτή η νέα πρόταση. Εμεί μελετάμε αυτή τη στιγμή μια νέα πρόταση, αναλύουμε την κατάσταση, Εμείς μελεταμε αυτη τη στιγμη μια νεα προταση αναλυουμε την κατασταση βασιζομαστε σε πιο πρόσφατα στοιχεία και μαζί με τη συνάδελφο κυρία Τάισεν μελετάμε το ζήτημα αυτό. Η συνάδελφός μου ασχολείται με την απασχόληση, με το τύχη της απασχόλησης. Ε, προφανώς θα συνεργαστούμε και με τον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμανς και με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης αφού το ζήτημα αφορά και τον κοινωνικό διάλογο και την εργασία. Είναι πολύ σαφές αυτό. Τώρα, δεν θέλω να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για να το πω ρεαλιστικά, στο δεύτερο εξάμεινο αυτού του έτους πιστεύω θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια πρόταση. η οποία βέβαια θα πρέπει να την οποία θα πρέπει να υποβάλουμε σε κάποια εκτίμηση επιπτώσεων. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ακούσατε τα πολυάριθμα συμπεράσματά μου. Εγώ προσδοκώ να συνεργαστώ μαζί σα και είδα ότι και εσεί έχετε μεγάλη βούληση για να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή είναι η νομοθεσία. Θα πρέπει πραγματικά να οδηγήσει σε μια κοινή αλλαγή. όχι μόνο για την πιο σημαντική πτυχή το να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών και των μητέρων στην Ευρώπη. Δεν χρειαζόμαστε κανόνε μόνο για τι γυναίκε. Χρειαζόμαστε κανόνε και για την Ευρώπη και για την ανάπτυξή τη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σα. Εκ μέρου του Συμβουλίου, καλούμε να πάρει το λόγο την κυρία Καλνίνα Λουκατσέβιτσα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. <clears throat> Πολλέ επικρίσει ε, ακούστηκαν σε σχέση με το Συμβούλιο απόψε Διαφωνώ με αυτές τις επικρίσεις. <clears throat> Για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να δώσουμε υποστήριξη σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Η απουσία υποστήριξης για την τρέχουσα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως απουσία βούλησης να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων γονέων. Και ως εκπρόσωπος ουσιαστικά ενός κράτους μέλους που προσφέρει γενναιόδορη ε, αμοιβή στις ε, γονεϊκές ε, άδειες μητρότητας και πατρότητας όπου μπορούν οι γονείς να επιλέξουν ο πατέρας ή η μητέρα το καθεστώς αυτό το οποίο θα επιλεγεί και να παραμείνουν για 18 μήνες για παράδειγμα οι μητέρες στο σπίτι τους Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι έχουμε στεναρή βούληση να παραμείνουμε πιστοί σε αυτές τις αρχές. Αυτό το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα είναι η απουσία υποστήριξης για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ως πρόταση που παρουσιάζεται από το Συμβούλιο για να μην υπερδραματοποιούμε την κατάσταση. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει μια νέα καλύτερη πρόταση. Αυτό θα ήταν πιο ρεαλιστικό και πιο επικαιροποιημένο. Θέλω να δραχθώ της ευκαιρίας να ευχαριστήσω να ευχαριστήσω την κυρία Κοράτσα Μπίρτ και την κυρία Σατία για τις ε, παρεμβάσεις τους ε, και τις ε, τοποθετήσεις τους ώστε να υπάρξει ένα νέο σύγχρονο σύστημα μητρικό, άδειας μητρότητας και να μην δακτυλοδεικτούμε και ποιοι είναι τάχα μου υπεύθυνοι για την απουσία λύσης. Ουσιαστικά κατανοεί πολύ καλά τη σπουδαιότητα της άδειας μητρότητας για τις ευρωπαϊκές οικογένειες στο Συμβούλιο η άδεια μητρότητα δεν πρέπει μεμονωμένα, απομονωμένα να εξετάζεται. Άλλα μέτρα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, το δικαίωμα σε υπηρεσίες και προσπελασιμότητα σε σχέση με ένα καθεστώ άδεια μητρότητα και την καλύτερη, τον καλύτερο επιμερισμό βαρών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ελαστικές, ελαστικές και ευέλικτες ρυθμίσεις που και αυτές διαδραματίζουν ένα ρόλο στι σύγχρονε κοινωνίε. Πολλέ μας. Πολλές ιδέες που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρα και να μας εμπνεύσουν σε αυτή την προσπάθεια το να γεννήσει μια γυναίκα ένα παιδί χρειάζεται η ίδια η γυναίκα και ο άνδρας της. Γιατί να κάνουμε λόγο λοιπόν μόνο για άδεια μητρότητας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Με ανησυχεί η ρητορική τοποθέτηση από διαφόρους μέσα στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων. Και οι άνδρες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα όπως και οι γυναίκες να συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών τους. Θα ήθελα λοιπόν να δραχθούμε αυτής της ευκαιρίας και να προσκαλέσω την ε, Επίτροπο, την κυρία Επίτροπο, προετοιμάζοντας μια νέα πρόταση, να προετοιμάσει μια σύγχρονη, επικαιροποιημένη πρόταση, όπου και οι δύο γονείς θα μπορούν να δραχθούν τις ευκαιρίες και να κάνουν χρήση υπέρ των παιδιών τους αυτή της άδεια. Πατρότητας, μητρότητας. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο είναι συνομοθέτης και η γνώμη του για την τρέχουσα πρόταση είναι σαφής εξ ου και πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Μπορούμε να συνεχίσουμε να διαφωνούμε επί της ε, ε, ενισχύ νομοθετικής πρότασης όπως έχει προταθεί και για άλλο χρονικό διάστημα ή μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με βάση μια νέα πρόταση. Το Συμβούλιο έχει κάνει την επιλογή του. Προσβλέπουμε τώρα στο να υπάρξει μια συμφωνία που θα καταστεί εφικτή στο άμεσο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Πιστεύω ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να συνεισφέρουν προς την θετική εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτό το σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η συζήτηση έληξε τώρα. Έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος.